Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Συνεχίζεται η διακοπή την 5η 21η ε, Μαΐου συνεδρίαση. Πριν περάσω στην έγκριση των πρακτικών θα ήθελα να ενημερώσω τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο όπως επίσης και τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα θεωρία